Βαρόνι Λάτφορντ, καταρχάς, έχετε πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω ότι αυτές οι δύο προφορικές ερωτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν στη... το Δεκέμβριο πέρσι ε, τις έχουν προλάβει τα γεγονότα. Αλλά και πάλι ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικονομικά δικαιώματα θα έχουν επιστρέψει πλέον μετά από απουσία αρκετών ετών και να ζητήσουμε να αποτελέσει προτεραιότητα το πρόγραμμα αυτό. Συνεχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία δεκαετία ζητά τα δικονομικά δικαιώματα ε, να λάβουν τη δέουσα προσοχή και δεν έχει ληφθεί δράση προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών στις ποινικέ διαδικασίες. Εμείς το έχουμε υποστηρίξει διότι ε, συλλαμβάνονται εγκληματίες και αυτοί που ε, απορρίπτουν το ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης είναι αυτοί οι οποίοι προάγουν τη μαφία και τους τρομοκράτες το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε και δικονομικέ εγγυήσει για να έχουμε απλουστευμένε ε, ποινικέ διαδικασίε διαμεθοριακά. Δεν θέλουν κάποιοι να αναλυφθεί δράση ε, για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Θέλουν να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψη μείων. Σε ορισμένε περιπτώσει είχαμε άρνηση δικαιοσύνη διότι δεν υπήρχε ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, η οποία να πηγαίνει συνάμα με την αμοιβαία αναγνώριση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ε, σε προφυλάκηση σε έξι μήνες για ανθρωποκτονία και δυστυχώς είναι θύμα ε, Λανθασμένη ταυτότητα και εδώ θεωρώ ότι έχει γίνει κακή χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Όταν συμφωνήθηκε το ένταλμα αυτό το 2002 υπήρχε κατανόηση από όλε τι πλευρέ ότι θα γίνεται αποτελεσματική του χρήση για να έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σε μια άλλη ε, χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα θα διασφαλίζονται συγκεκριμένα ε, δικαιώματα και δεν θα υπάρχει κακοδικία. Πολλά κράτη-μέλη έχουν παραβιάσει αυτό το δικαίωμα και έχει απορριφθεί και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για μία απόφαση για, τα ποινικά, για τις ποινικέ διαδικασίες και αυτή τη στιγμή αυτό που λαμβάνουμε είναι το καλύτερο που μπορούμε να λάβουμε. Είμαι ευγνώμων που το ξαναξεκίνησε το θέμα η Σουηδική Προεδρία, αλλά αποτελεί έναν οδικό χάρτη και μόνον για μια βαθμιδόν διαδικασία. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο υπόσχεται μόνο να το σκεφτεί και να μην ε, νομοθετήσει για το θέμα της... Ε, για τις ποινές με αναστολή. Θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τα δικαστήρια στις άλλες χώρες μέλη και δυστυχώς υπάρχουν μεγαλύτερες επικρίσεις και θα υπάρχουν λεώνα και περισσότερες επικρίσεις αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εγγύσεις για τα ποινικά δικαιώματα και δεν μας ενδιαφέρουν ε, μόνο τα θέματα για τους πολίτες που δεν έχουν κατάλληλες διασφαλίσεις και κατάλληλα δικαιώματα. Τα θέματα αυτά αφορούν και τους δικαστές αλλά και για τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούν να διεξάγουν σωστά το έργο τους. Πιστεύω ότι η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Άντελμα Σύλληψη θα πρέπει να είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την έκδοση κάποιου, ε, παρά το γεγονό ότι στο Συμβούλιο μπορεί να μην αρέσει κάτι τέτοιο. Κατά την εφαρμογή του μέτρου λέγεται ότι ε, δεν γίνεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα το δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ορισμένες φορές ε, χρησιμοποιεί το επιχείρημα αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ε, και λένε κάποιοι ότι δεν χρειάζονται να ληφθούν ευρωπαϊκά μέτρα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σεβασμό σε κάποια κράτη-μέλη και πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγουν στο δικαστήριο στο Στρασβούργο ακριβώς για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή η ε, νομοθεσία ε, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δεχτούν ε, κάποιους κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να γίνει εφαρμογή των κανονών και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν διαδικασίες επιπαραβάση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα υποπτεύει τις διαδικασίες. Τα μέτρα λοιπόν θα πρέπει να συνάδουν με τα όσα έχουμε αποφασίσει, να μην τα υποσκάπτουν και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη εφαρμογή τους. Άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στη διερμηνία και στη μετάφραση σε μία δίκη, όπως ε, ε, συμφωνήθηκε στην απόφαση πλαίσιο του 2009, δεν είναι τόσο φιλόδοξο όσο είχαμε αρχικά. Επομένως, το πρώτο μέτρο θεωρούμε ότι δεν είναι όσο το δυνατόν υψηλέτερο επίπεδο γίνεται. Ελπίζω να έχουμε καλύτερα ε, αποτελέσματα στο επόμενο στάδιο των ε, δικονομικών δικαιωμάτων. Τα θέματα της μετάφρασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλα μέτρα όπως το δικαίωμα στην, σε συνήγορο, ε, καλή επικοινωνία με το δικαστήριο και ούτω καθεξής. Ε, ελπίζω λοιπόν το δικό χάρτης να προχωρήσει αρκετά γρήγορα ώστε να έχουμε ένα καλό ε, αποτέλεσμα και δικαίωμα στη η δίκη, κάτι το οποίο περιμένουμε εδώ και καιρό. Για το Συμβούλιο ο κύριο Λόπες Γκαγίδο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε αυτή την ερώτηση κυρία Λάτφορτ, και για την παρέμβασή σας. Την ε, πρόταση παρουσιάζουν επίσης και η κυρία Αντωνέσκου, Ρομέρο Λόπες, Ζαουτάλα και Ταβάρες. Όντως πρόκειται για ένα θέμα μεγίστη σημασίας όπως είναι τα δικοδονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Και Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με την αξιολόγηση και τη σημασία που προσδίδεται στο θέμα αυτό, όπως είπατε κι εσείς, και επίσης συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς στην ερώτησή σας λέτε ότι η Σουηδική Προεδρία έκανε μια σημαντική πρόοδο. Όντως η Σουηδική Προεδρία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς ε, το θέμα αυτό συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο ένα γενικό προσανατολισμός για το δικαίωμα στη μετάφραση και στη διερμηνία στις ε, ποινικέ διαδικασίε. και το Νοέμβριο το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα σχέδιο προκειμένου να προχωρήσουν ε, κάποια επιπλέον μέτρα, όπως ζήτησε η κυρία Λάτφορντ, και να έχουμε επιπλέον μέτρα για τις ποινικέ διαδικασίες και τα δικονομικά δικαιώματα το δικαίωμα στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση για τα δικαιώματα ε, του καθενός, καθώς επίσης και τα ε, καθήκοντα που έχει κάποιος σε μια ποινική διαδικασία, στην, ε, στο δικαίωμα σε νομική συνδρομή, στην επικοινωνία με την οικογένειά τους, με προξενικές αρχές και τις ειδικέ εγγυήσεις που πρέπει να δίνονται σε θέματα προστασίας για κατηγορημένους οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Αυτά λοιπόν τιμήθησαν στο Συμβούλιο επί Σουηδικής Προεδρίας. Εσείς στη συνέχεια λέτε, καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχει κάποια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συνεχίσει αυτή η εργασία ως προτεραιότητα. Και εδώ σας απαντούμε, ναι, πρόκειται για προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε προς αυτή την άγουσα. Με τι, με τι κατευθύνσεις η Ισπανική Προεδρία αυτό που θα κάνει είναι να προσπαθήσει να υιοθετηθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οδηγία που ξεκίνησαν τρία κράτη-μέλη για τα δικαίωμα στη διερμηνία και στη μετάφραση στις ποινικέ διαδικασίε. Δεν υπήρξε δυνατότητα να συνεχιστεί η πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρία κράτη-μέλη αντικατέστησαν αυτή την πρωτοβουλία και θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία να εγκριθεί σε συνεργασία πάντα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επιπλέον Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στα ε, δικονομικά δικαιώματα να προχωρήσει τα θέματα αυτά και είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να μπορέσουμε ε, από κοινού Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα εγκρίνουμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να σας πω ότι η Ισπανική Προεδρία έχει προβλέψει ένα σεμινάριο στη Μαδρίτη το Μάρτιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαιωμάτων ε, και το θέμα είναι δικονομικά δικαιώματα και συγκεκριμένε. Ε, συγκεκριμένα πρότυπα επί του θέματος. Και αυτό σας δείχνει πόσο συμμερεζόμαστε από κοινού μαζί σας και με όσους ε, προσυπογράφουν αυτή την ερώτηση το κατεπήγον του θέματος που ότι πρέπει να ρυθμιστεί, πρέπει να εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά θα ενημερώνουμε συνεχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, πρόοδο των εργασιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μπαρό. Κυρία Λάτφορντ, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Γνωρίζετε πόση σημασία αποδίδω σε αυτές τις οικονομικές εγγύσεις. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγωνίζεται για ελάχιστους κοινούς κανόνες σε θέματα υπεράσπισης. για να γενικευθούν αυτά σε όλες τις ποινικέ διαδικασίες στην Ευρώπη. Αυτό είναι απαραίτητο για την δικαστική συνεργασία. Είναι η προϋπόθεση, η προϋπόθεση για την αμοιβαία εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε πολλές προσπάθειες για την θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, χάρη στη Σουηδική Προεδρία εγκρίθηκε ο δικός χάρτης από το Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2009. Αυτό είναι ένα σημαντικό σταθμό για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα δικονομικά δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη με την πράξη αυτή συμφώνησαν ως προς το πεδίο εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας και για την ανάγκη θέσπισής της με απόλυτη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άκουσα όπως και εσείς αυτά που μας είπε ο Υπουργός Λόπες Γκαρίγκο που μας εξήγησε σαφώς τι προτίθεται να κάνει η Ισπανική Προεδρία ώστε να θεσπιστούν αυτά τα πρώτα μέτρα που θα μας οδηγήσουν σε ένα φάσμα ελάχιστων βασικών εγγύσεων. Η έγκριση του οδικού χάρτη αποδείχθηκε μια σωστή λύση. Αυτή η προσέγγιση θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο. Η βήμα προς βήμα, η step by step διαδικασία σημαίνει όχι μόνο ότι κάθε δικαίωμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης ανάλυσης στα πλαίσια της νομοθετικής πρότασης, αλλά επίσης ότι στη διαπραγμάτευση κάθε δικαίωμα μπορεί να εξετάζεται μεμονωμένα έτσι ώστε να αποφευθούν τα παζαρέματα που καμιά φορά χαρακτηρίζουν τα νομοθετικά κείμενα τα οποία παρά είναι σφαιρικά και γενικά επιτρέποντας έτσι σε κάποια κράτη-μέλη να θέσουν σε ε, ομοιρία την διαπραγμάτευση για να εξασφαλίσουν κάποιο πλεονέκτημα για ένα συγκεκριμένο σημείο. Κυρία Λάτφορντ, η νέα Επιτροπή, είμαι βέβαιος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποβάλει όλες τις νομιθετικές ε, προτάσεις που προβλέπουν στον οδικό χάρτη ώστε να θεσπιστούν το νωρίτερο δυνατό. Τώρα, στο δικαίωμα ε, σε διερμηνία και μετάφραση, το πρώτο μέτρο που προβλέπει ο δικός χάρτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε γνώση της πρωτοβουλίας που ανέλαβαν αρκετά κράτη-μέλη. Αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται, πρέπει να σας πω, στην πρόταση της Επιτροπής του Ιουλίου 2009 και στις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα το δεύτερο εξάμεινο του 2009 σε επίπεδο Συμβουλίου. Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία των κρατών μελών, ωστόσο, δεν συμβαδίζει απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με την ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Η παλαιότερη πρόταση της Επιτροπής που έκανε υποχρεωτική την ε, ε, διερμηνία των, στις συναντήσεις μεταξύ ε, δικηγόρου και κατηγορουμένου δεν τηρείται απόλυτα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των κρατών μελών που περιορίζει αυτό το δικαίωμα στην επικοινωνία που γίνεται στην παρουσία των αστυνομικών αρχών και στη διάρκεια της δίκης. Η παλαιά πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε επίσης δικαίωμα σε μετάφραση, ένα δικαίωμα πιο πλήρες σε αυτό το κείμενο της Επιτροπής. Αλλά βεβαίως θα χρειαστεί να γίνει δουλειά μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα φιλόδοξο κείμενο για τα δικονομικά δικαιώματα, κάτι το απαραίτητο. θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά έναν ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, χώρο δικαιοσύνης, ένα κείμενο το οποίο θα τηρεί τα πρότυπα και, τους, θα τα τηρεί τα πρότυπα που έχει θέσει η ΕΣΔΑ και η νομολογία του Ευρωπαϊκού του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είμαι βέβαιος θα μπορέσουμε να στηριχθούμε στην δράση σε αυτόν τον τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακόμα μια φορά ε, θέλω να πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσει και όλη την απαιτούμενη βοήθεια η Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο και τώρα κύριος Νατανέσκου για δύο λεπτά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Παρόλο που υπάρχει σαφής πρόοδος όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων και αυτό έχει καταγραφεί και την ίδια ώρα βλέπουμε δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος στα δικαιώματα των κατηγορουμένων τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθότι σήμερα βλέπουμε ότι έχουν υποχωρήσει τα δικαιώματα αυτά στις ποινικέ διαδικασίες, τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Η Σουηδική Προεδρία λοιπόν ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει αυτόν τον ε, οδικό χάρτη, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, όπως επίσης το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας για τους ε, κατηγορούμενους. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό που προβλέπει και η Συμφωνία της Λισαβόνας και εμείς θα πρέπει να εκφράσουμε εδώ την ανησυχία μας για το θέμα των δικαιωμάτων και θέλουμε να θέσουμε το θέμα αυτό πολύ σοβαρά στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. 13 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, υπέβαλαν μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ελπίζουμε να βελτιωθεί το αρχικό κείμενο όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται σε μια τέτοια διαδικασία, ιδιαίτερα το δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνία. Η εγγύηση της πρόσβασης σε μια υπεράσπιση σε σωστή ενημέρωση, ιδιαίτερα όσον αφορά ενημέρωση για τα δικαιώματά τους. Οι προτάσεις αυτές θα υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν και πιστεύω ότι σήμερα ενώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει οπωσδήποτε να ιθωτηθούν κοινά πρότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρομέρο Λόπες για δύο λεπτά. Καταρχάς να χαιρετήσω την Ισπανική Προεδρία και ταυτόχρονα να τονίσω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι η πρώτη πρωτοβουλία για τα δικονομικά δικαιώματα ένα θέμα το οποίο συζητούσαμε και ε, που επανέφερε στη συζήτηση η Σουηδική Προεδρία. Αυτή η πρόταση πρωτοβουλίας έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική έδρα και έχει γίνει και μια πρώτη συζήτηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρη η ερώτηση λόγω της σημασίας του θέματος. Σαφώς ε, χρήζει μεγάλες βελτίωσεις και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι αλήθεια ότι όπως είπε και ο κύριος Μπαρό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ πιο φιλόδοξη γι' αυτό και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το κατόφλι. Είναι ένα κατόφλι το οποίο έχει μια μακρά πορεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούν ε, με την αντίσταση των κρατών μελών. Τη Σουηδική Προεδρία με τον οδικό χάρτη έκανε μία απόπειρα να ξεπλοκάρει το ζήτημα, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη για τα κράτη-μέλη. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει αλλάξει η κατάσταση διότι πλέον το Κοινοβούλιο αποφασίζει και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να δουν αυτά τα δικονομικά δικαιώματα υπό ένα νέο πρίσμα και αυτό ζητάμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε αυτά τα δικονομικά δικαιώματα λοιπόν να συζητηθούν σε ένα πακέτο να αναγνωριστεί το δικαίωμα στη μετάφραση και στη διερμηνία αλλά να μην ξεχνάμε και το δικαίωμα στην νομική συνδρομή και στις πληροφορίες. Ε, κάθε χρόνο προχωράει το θέμα αντί για αυτό να ε, περνάνε ε, κάθε χρόνο να παρουσιάζεται και από ένα νέο δικαίωμα θα πρέπει να συνθεθούν όλα αυτά τα πράγματα και να παρουσιαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις αλλά αν θέλουμε να έχουμε ένα χώρο δικαιοσύνης και ελευθερίας θα πρέπει να προάγουμε τις αξίες μας και να τις μεταλαμπαδεύσουμε και στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βότσον για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο πρότεινε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2001 το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ακόμα υπάρχει ψηλά σε ένα ράφι αυτό το ένταλμα και ξέρετε ότι ο κύριος Μπιν Λάντερ μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτό που σημαίνει αυτή η πρόταση. Τότε θυμάμαι, είχαμε επιμείνει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εγγύησης και δικονομικά δικαιώματα. Το 2002 έγιναν οι πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ταχεία διαδικασία. Γιατί όμως παραμένει το θέμα αυτό εγκλωβισμένο στους μεάνδρους του Συμβουλίου, ενώ έχουν ε, εγκριθεί κάποιες προτάσεις. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης έχει αντικαταστήσει τη διαδικασία της ε, απέλασης. Υπάρχουν άμεσες επαφές και της έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί να μην επιταχύνουμε τη διαδικασία, καθότι υπάρχουν θέματα που αφορούν υπηκός των κρατών μελών και αφορούν όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Υπάρχει η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην οποία βασίζονται αυτές οι διαδικασίες. Και σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες αν αμφιβάλλουν αν τα θέματα αυτά θα προχωρήσουν. Σήμερα υπάρχουν Βρετανοί υπήκοοι οι οποίοι βρίσκονται στην Ουγγαρία και περιμένουν τη δίκη τους. Η σύλληψή τους και η φυλάκισή τους έγινε πριν από μήνες. Ο ένας έχει ήδη χάσει τη δουλειά του, η οικογένειά του δεν έχει πλέον ε, εισοδήματα. Θα μπορούσαν να ήταν αθώοι αυτοί οι άνθρωποι για τα εγκλήματα οποία τους κατηγορούν. Και βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά χαλάει τελείως η εικόνα και δυσφημίζεται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν επίγον το θέμα και θα πρέπει να επιληφθούμε το συντομότερο δυνατόν. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι είσαστε και ο νονός αυτού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χαουτάλα για τρία λεπτά όμως. Yes, he was waving it. Do you accept Αναφέρθηκε ο Μπιν Λάντεν και τα γεγονότα της 9 Σεπτεμβρίου σαν ε, το κινητήρια δύναμη για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εναντίον δολοφόνων και τρομοκρατών και άλλων υπέτειων βαρύτατων εγκλημάτων. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε, δεν χρησιμοποίησα δικαιολογία των Μπιν Λάντεν. Είπα ότι μας βοήθησε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Είχε σκοπό να καταπολεμήσει όλα τα βαριά εγκλήματα, όχι μόνο τις τρομοκρατικές ενέργειες. Εκείνους οι οποίοι καταπατούν το κράτος δικαίω στην Ήπειρό μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψης ώστε να εξασφαλίσουμε τη δέουσα προστασία στου Ευρωπαίου πολίτε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Βοτσακόφσκι για ένα λεπτά. I'm sorry, forgive me. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, έπρεπε να δώσω το λόγο πριν στην κυρία Χάουταλα. Ζητώ συγγνώμη κυρία Χάουταλα. Δεν πειράζει κύριε Πρόεδρε. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το να ισχύουν ορισμένα κριτήρια και ελάχιστε εγγυήσει για τις δικονομικέ διαδικασίες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψη. Σε ορισμένε χώρες το ένταλμα σύλληψη έχει χτιστεί πάνω στην άμμο. Έχει χτιστεί πάνω στην άμμο διότι με βάση την παραδοχή ότι έχουμε εμπιστοσύνη μεν στους δε και στα ε, συστήματα ποινική δικαιοσύνη ότι τα δικαιώματα των πολιτών γίνονται σεβαστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Όπω είπαν συνάδελφοι προηγουμένω, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μπορούσα να σα διηγηθώ πάρα πολλέ ιστορίε που δείχνουν ότι δεν συνισχύει αυτό και γι' αυτό επήγει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπε ο συνάδελφο. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα στηρίζεται σε ελάχιστε εγγυήσει και μα δίνει αυτή την ευκαιρία η συνδίκη τη Λισαβόνα. Διότι πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλήρε νομοθετικέ εξουσίε όπως και το Συμβούλιο, παράλληλα με το Συμβούλιο. Και με τα χαράς άκουσα τον Επίτροπο να μας λέει ότι έχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη συνεργασία. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν προκειμένου να δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα και να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις των κρατών μελών. Θα μπορούσα να σας διηγηθώ ιστορίες που δεν γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου, παρόλο που χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Στη Φιλανδία υπάρχει ένα ζευγάρι που είναι κρατούμενοι, ο Άσιακα και Μάλι Κατάγεφ, που ήρθαν από τη Λιθουανία, όπου επί χρόνια ε, λειτουργούσαν ένα ορφανοτροφείο. Ξαφνικά στην Τσετσενία για παιδιά από την Τσετσενία παρενέβη στη δραστηριότητά τους η αστυνομία της Τσετσενίας ξαφνικά με την δικαιολογία ότι υπήρχαν φαινόμενα οικογενειακής βίας. Ε, το ζευγάρι αυτό ε, ε, βρίσκεται τώρα στη Φιλανδία, η Λιθουανία ζητά την έκδοσή του. Ε, την επόμενη εβδομάδα στο Ελσίνκι. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Η Φιλανδία χρειάζεται να, πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι το ζευγάρι αυτό θα δικαστεί με δίκαιο τρόπο στη Λιθουανία, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει βεβαιότητα. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα αποτυχίας ή ατελούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς για να υπάρξει απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των κρατών μελών για την σωστή εφαρμογή της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αουτάλα. Ένας νέος Πολωνός καταδικάστηκε για βιασμό στη Μεγάλη Βρετανία σαν αποτέλεσμα δημοσιευμάτων στον τύπο. Η διαδικασία δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε και σήμερα κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ποινή θανάτου παρόλο που στην Πολωνία για αυτό το έγκλημα η ποινή είναι 12 ετής φυλάκιση και όχι ποινή θανάτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το παράδειγμα σας δείχνει ότι τα διαφορετικά συστήματα οδηγούν σε αυτές τις ε, στρεβλώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκτέλεση των ποινών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εδώ μια κοινή αντιμετώπιση, κοινά πρότυπα, καθότι σε μια χώρα μπορεί η κατάσταση να είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό και εγώ στηρίζω τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχουμε τα κράτη-μέλη και έχουμε και τους πολίτες που εδώ εκπροσωπούνται από το ερωτώμα σώμα. Πολύ συχνά, έχοντας διαπιστώσει και οι δύο σώμασοι τι προβλήματα υπάρχουν και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τα διάφορα δικαστικά συστήματα, ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτή είναι μία από τις κλασικές περιπτώσεις. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, επιταχύνει τις ε, διαδικασίες, ε, διευκολύνει τα δικαστικά συστήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνία, και εγώ ασχολήθηκα με όλα αυτά τα θέματα με τη συνάδελφο Λάτφορντ και αυτά είναι ουσιαστικά, διότι ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη όταν υπάρχουν ε, τέτοια δικαστικά θέματα σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο να παρουσιάσουν ένα κείμενο το οποίο χάρη στη διαδικασία της συναπόφασης θα μας βοηθήσει να φέρουμε σε αίσιο τέλος το θέμα των δικονομικών δικαιωμάτων. Έχουμε δύο άτομα από την περιφέρειά μου, το Μάικολ Τέρνερ που και έναν ακόμα που βρίσκονται σε μια κεντρική φυλακή στη Βουδαπέστη. Είναι ε, προφυλακισμένοι από τις 3 Δεκεμβρίου, ε, περιμένουν τη δίκη, δεν έχει ακόμα καθυραστεί η ημερομηνία της δίκης και ε, οι συνθήκες φυλάκισής τους είναι πολύ δύσκολες, δεν έχουν επαφή ο ένας με τον άλλον, βρίσκονται σε ένα κελί με άλλους τρεις φυλακισμένους και είναι σε περιορισμό στο κελί όλη την ημέρα, δικαιούνται τρία τηλεφωνήματα και ένα ντού την εβδομάδα και δικαιούνται και μία επίσκεψη ε, μέλους της οικογένειάς τους μία φορά την εβδομάδα. Ουσιαστικά βρίσκονται σε απομόνωση. Το πρόβλημα της γλώσσας ε, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο αυτή την απομόνωση. Κατηγορούνται για κάποιο μικροαδίκημα, δεν είναι δολοφόνοι και βρίσκονται στην ε, ε, φυλακή λόγω του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ουσιαστικά με μια ε, εξαφάνισε όλα τα δικαιώματα που έχουν καθοριστεί στη Βρετανία μέσα σε χίλια χρόνια. Μην κουνάτε έτσι το κεφάλι σας κύριε Βότσον, θα πρέπει να ζητάτε συγγνώμη. Η λανθασμένη ταυτότητα και η κλοπή ταυτότητας σημαίνει ότι αυτό που συνέβη στον Τζέισον και στον Μάικολ μπορεί να συμβεί κάλλιστα και σε οποιονδήποτε άλλο Βρετανό πολίτη ανα πάσα στιγμή το Εργατικό Κόμμα και το Συντηρητικό κόμμα, όλα αυτά τα κόμματα υπερψήφισαν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Για να παραφράσω το Ζολά, Κατηγορώ και εγώ, κατηγορώ τα κόμματα του Βρετανικού πολιτικού συστήματος, διότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και την υποστήριξή τους. Κάθε Βρετανός λοιπόν κινδυνεύει να συλληφθεί τυχαία. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, eh, magyar emberként és büntetőjogászként szégyelnem. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σαν ειδικό του ποινικού δικαίου να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται σε περιπτώσεις, σε υποθέσεις στην Ουγγαρία δύο ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές ομάδες αναφέρθηκαν σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά που λέτε για τη χώρα μου. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας ζητήσω και όλους εσάς που είστε εδώ τόσο αργά σε αυτή τη συζήτηση στην υπόθεση αυτή ξένων ε, υπηκών οι οποίοι πραγματικά υποβάλλονται σε τέτοιες παραβιάσεις των δικονομικών τους δικαιωμάτων στην Ουγγαρία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως και οι παρόμοιες περιπτώσεις Ούγγρων οι οποίοι κρατούνται τους τελευταίους εννέα μήνες και οι οποίοι υποβάλλονται σε πιέσεις και κατηγορούνται για τρομοκρατικές πράξεις. Δεν μπορεί όμως να αποδειχτεί τίποτα οι Ουγγρικές αρχές δεν μπορούν να αποδείξουν αυτές τις κατηγορίες, είναι απομονωμένοι, δεν μπορούν να έχουν σε επαφή με τις οικογένειές τους ή με άλλους. Γι' αυτό και θα ήθελα πραγματικά από κοινού να βοηθήσουμε ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ουγγαρία και να αποφευχθούν οι καταχρήσεις και οι παραβιάσεις αυτών των δικονομικών δικαιωμάτων και η έλλειψη εγγυήσεων στην Ουγγαρία. ένα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Λόπες, ο κύριος Λόπες Γκαρίγκο δεν θα ενοχληθεί αν αναφερθώ πρώτα στον κύριο Μπαρό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε με εκείνον πάλι ξανά σε αυτή την αίθουσα και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες, για όλο το αίσθημα συνεργασίας που επέδειξε πάντα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα των δικονομικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να προσθέσω και τη δική μου φωνή σε εκείνους που πριν από μένα είπαν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη της ασφάλειας αλλά και μια Ευρώπη της δικαιοσύνης παράλληλα. Όλες οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται ε, στα δικανομικά δικαιώματα είναι λοιπόν ύψης της σημασίας. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να βοηθήσουμε τα θύματα για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών που προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που απευθύνουμε λοιπόν στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σωστά είπε ο Βότσον πριν από μένα. Δεν, δεν είναι σωστό μετά από 8 χρόνια να έχουμε ασχοληθεί μόνο με μία πτυχή του προβλήματος. Πρέπει λοιπόν να ενεργήσουμε πλέον από εδώ και πέρα ταχύτερα αυτή είναι μια υποχρέωση που ανήκει στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω κύριε Μπαρό ότι η επόμενη Επιτροπή θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες ε, σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα και δεν θα περιοριστεί μόνο στο θέμα της μετάφρασης και της διερμηνίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπένοβα, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα δικονομικά δικαιώματα σε αυτές τις ποινικέ διαδικασίες είναι ένα ουσιαστικό θέμα όταν μιλάμε για την ασφάλεια του δικαίου. Και πιστεύω ότι πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν, ιδιαίτερα το δικαίωμα για μετάφραση, για δικαίωμα επικοινωνίας, επαφής με τις ε, προξενικές αρχές και υπεράσπισης. Αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να τα προασπίσουμε, να υπάρξουν κοινά πρότυπα, γιατί βεβαίως πρόκειται, όπως σας είπα, για θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Η συμμετοχή μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προϋποθέτει την προάσπιση αυτών των δικονομικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η συμμετοχή στην ποινική διαδικασία και των κατηγορουμένων και των θυμάτων θα πρέπει να γίνεται βάσει κοινών προτύπων, βάσει δημοκρατικών διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούνται. Αυτός είναι και ο στόχος που θα πρέπει εμείς εδώ να προασπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πέρκμαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ καλούμε το Συμβούλιο να συνεχίσει την προάσπιση των δικονομικών δικαιωμάτων στις ποινικέ διαδικασίες. Υπάρχει μια κοινή διαδικασία, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που ουσιαστικά αποτελεί την ασφαλιστική δικλίδα και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι κάποιες από τις εγγύσεις έχουν καταργηθεί βλέπουμε ότι ο Άντριου Σίνιορ, παραδείγματο χάρη, υπήκος τη χώρα μου και τη εκλογική μου επικράτεια, έχει εκδοθεί χωρίς να μπορέσει απολύτω κανένα αγγλικό δικαστήριο, βρετανικό δικαστήριο, να προλάβει και να αποφύγει αυτή την άδικη έκδοσή του. Πρόκειται πλέον για μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Όταν μιλάμε για την έκδοση βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ατόμων που δεν υποβάλλονται σήμερα σε δίκαιη δίκη. Όπως ο κύριος Σίμονς, ο οποίος βρίσκεται στον Κορυδαλό. Βεβαίως, ακούμε σήμερα πολλούς οι οποίοι λυπούνται, πολύ αργά όμως, και κροκοδίλια δάκρυα για την περίπτωση του κυρίου αυτού. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι υποχωρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και υποβαθμίζονται. Εάν θέλουμε αυστηρά πρότυπα στην Ευρώπη για τις ποινικέ διαδικασίες, θα πρέπει οι διατάξεις της Μάγνα Κάρτα να υιοθετηθούν και να γίνουν οι κοινέ ευρωπαϊκές εγγύσεις και πρότυπα. Ξεκινάει η διαδικασία Catch Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Είναι καθοριστικό να προωθήσουμε κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία απόδοσης ποινικών ευθυνών όπως συζητάμε μέχρι τώρα. η έννοια κλειδί είναι η έννοια της εμπιστοσύνης. θέλουμε εμπιστοσύνη του ευρωπαίου πολίτη που βρίσκεται ενώπιον στη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. θέλουμε επίσης εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη συνεργασία τους και την απονομή της δικαιοσύνης τελικά σε κάθε ένα που ε, καλείται να λογοδοτήσει σε αυτή. ένα τελευταίο που θέλω να επισημάνω χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη από όλους μας σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης και όσο δεν προωθούμε τα κοινά αυτά πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλώς ή κακώς κάποιες φορές θα υπάρχουν και κάποιοι εγκληματίες οι οποίοι θα αξιοποιούν τα κοινά που θα υπάρχουν και τελικά δεν θα έχουμε την απονομή δικαιοσύνης που επιδιώκουμε ακριβώς γιατί δεν θα υπάρχουν τα κοινά αυτά πλαίσια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το Συμβούλιο κύριος Λόπες ε, Γκάριδο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι διαπίστωσα από τις ε, παρεμβάσεις ε, πολλών από τους ευρωβουλευτές που ακούσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από πολύ διαφορετικές πολιτικές ομάδες, μία σύμπτωση απόψεων στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δικονομικά δικαιώματα. Να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκαιο για τα εγγυήσεις ε, στα δικονομικά δικαιώματα. Υπήρχε ταύτιση απόψεων ε, από όλους τους παρεμβαίνοντες ε, και από όλες τις πολιτικές ομάδες ώστε να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικονομικά δικαιώματα. Αυτό άλλωστε καταδεικνύει και πόσο σημαντική είναι η διαδικασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, η Ευρώπη των πολιτών, του ευρωπαϊκού χώρου, την ε, σημασία της εφαρμογής της Εθνικής της Λισαβόνας. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η Ισπανική Προεδρία στους επόμενους έξι μήνες και νομίζω ότι ε, έλαβε και μια διαφυρισβήτητη στήριξη σε όλες τις παρεμβάσεις που άκουσα ε, από διάφορα επιχειρήματα, διάφορες προοπτικές. Υπάρχει ανάγκη να έχουμε δικονομικά δικαιώματα εναρμονισμών. Ε, μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Μπένοβα. Αυτό γίνεται σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέει η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ολοκληρώνοντας να πω κύριε Πρόεδρε ότι το Συμβούλιο, η Ισπανική Προεδρία θα εργαστεί ώστε να τεθούν σε εφαρμογή όλες αυτές οι ε, εγγυήσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την οδηγία που ήδη έχει ξεκινήσει ε, κατόπιν πρωτοβουλία, ε, υπενθυμίζω, τριών κρατών μελών. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω κάτι για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Κάποιοι το επέκριναν. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη αποτελεί θεμελιώδες παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και τη συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να σας το πω φωναχτά από μια χώρα όπως η Ισπανία που ακόμα πλήττεται από την τρομοκρατία και για την οποία το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο κατά της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός έχει δίκιο και ο κύριος Κοέλλο πολύ σωστά είπε προηγουμένως Ευρώπη της ασφάλειας αλλά και Ευρώπη της δικαιοσύνης. Βεβαίως κύριε Βότσον, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ε, αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό. Αλλά είναι σωστό ότι παράλληλα το πρέπει να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Χώρος και να οργανωθεί και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε για την Ευρώπη της δικαιοσύνης με σκοπό να υπάρχει εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο απονέμε τη δικαιοσύνη παντού στην Ευρώπη. Και σχετικά θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τους συντάκτες της ερώτησης και να τονίσω και πάλι ότι με βάση το κείμενο που εκφράζει τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια βεβαίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ισπανικής Προεδρίας θα φροντίσει η ποιότητα του κειμένου να είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα του τωρινού κειμένου. Επίσης προσθέτω ότι θα φροντίσουμε σε έφετο χρόνο να διατυπώσουμε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις ώστε να μην απαιτηθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία από πλευρά των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται, ε, προετοιμάζει ήδη την πρόταση για τα δικαιώματα. Θα προσπαθήσει να εφαρμοστούν, να θεσπιστούν αυτά που προβλέπονται στον οδικό χάρτη το ταχύτερο δυνατό. Η διάρκεια του ενός έτους είναι ενδεικτική. Αν το επιτρέψουν οι διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι προφανές αυτό. Πάντως εγώ ακράδαντα πιστεύω ότι τα πνεύματα έχουν ερημάσει. Το πολιετές πρόγραμμα της Στοκχόλμης μας δημιουργεί μια ουσιαστική υποχρέωση να καταλήξουμε σύντομα σε αποτελέσματα και από τότε που ανέλαβα αυτές τις αρμοδιότητες πρέπει να σας πω ότι έκανα κάθε, προσπάθεια για να προχωρήσει αυτός ο φάκελος για τα δικονομικά δικαιώματα. Παρόλο που επιλέξαμε την ε, διαδικασία, ε, τη βήμα προς βήμα διαδικασία, step ε, by step, προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς και είμαι πεπισμένος ότι θα προοδεύσει πάρα πολύ η Ευρώπη της δικαιοσύνης το 2010. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ότι υπάρχουν πολλοί εκτός εθούσης που συμφωνούν με αυτά που είπε ε, ο κύριος Κοέλιο και σας ευχαριστούμε επίσης για όλη την βοήθεια και τη συνεργασία που είχαμε μαζί σας. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είναι η εμπορία ανθρώπων. Πρώτος ομιλητής η κυρία Αναχέντ για δυόμιση λεπτά.